Διαρευνητικέ συνομιλίες. Ωραία. Τι ωραία, τελειώσαμε και τις ερωτήσεις με μια ερώτηση για τον τουρισμό, έτσι με κάτι θετικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τις ερωτήσεις τους, πολλές και διάφορες, και να ευχαριστήσω και την υποψήφια Επιτροπό για τις απαντήσεις της ε, τώρα, κυρία η υποψηφία, αν μπορείτε σε πέντε λεπτά να κάνετε μία σύνοψη όσων θα θέλατε εσείς να τονίσετε από τη σημερινή ακρόαση τα πιο σημαντικά ζητήματα και μετά η Προεδρία της Ήτρε ε, ο κύριος Μπούζεκ θα κάνει κάποιες παρατηρήσεις και μετά θα σας ενημερώσω ε, για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Υποψήφια Επίτροπος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω πως η συζήτηση αυτή θα είναι η αρχή μιας καλής ε, συνεργασίας και ελπίζω να συνεχίσει συνεργασία στο πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τακτικού διαλόγου και θα σας ε, και θα δεσμευτώ ενώπιόν σας για το εξής. Θα είμαι στρατευμένη όσον αφορά την επίτευξη όλων των δυνατοτήτων της εσωτερικής αγοράς και θα καταβάλω άοκνες προσπάθειες για να λύσουμε τα διάφορα προβλήματα ένα-ένα και για να βρούμε αμοιβαία επαφελείς λύσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γνωρίζω την σημασία του Κοινοβουλίου και της εντολής του και βεβαίως θα είμαι υπόλογη σε εσά. Και βεβαίως ε, μετά από τις ερωτήσεις σας έχω την εντύπωση πως ε, το χαρτοφυλάκι αυτό είναι σημαντικό για όλες τις ομάδες παρά τις διαφορές που υπάρχουν και μας δίνει την δυνατότητα για ανάπτυξη και δουλειές. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ που επέζησα κιόλα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία υποψήφια επίτροπε για όλες τις απαντήσεις σας. και για τις καταληκτικές σας παρατηρήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στην ε, ε ακρόαση αυτή, τους ε, ακροατές από το διαδίκτυο και θα ήθελα στο τέλος της ακροασής μας να σας δώσω μια πληροφορία που δεν είχα το θάρρος να σας δώσω στην αρχή ότι προέρχομαι από την ίδια περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και η υποψήφια κυρία Επίτροπος. Είναι μια πολύ βιομηχανική περιοχή. Και χρειάστηκε να περάσουμε μια πολύ δύσκολη διαδικασία αναδιάρθρωσης όλου του βιομηχανικού ιστού της περιοχής αυτής. Έχει λοιπόν από αυτή την άποψη μεγάλη εμπειρία η κυρία υποψήφια τρόπος και συγχρόνως έχει μάθει πολλά και για το περιβάλλον που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει μια περιοχή που έχει ισχυρή χαλιβουργία και χημική βιομηχανία και έχει φυσικά και 7 χρόνια εμπειρία στην κυβέρνηση της Πολωνίας ως και αναπληρωτής πρωθυπουργός. και ελπίζω ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να έρθουμε σε επαφή μαζί της τα επόμενα πέντε χρόνια γιατί όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες μας. Και σας ευχαριστώ και πάλι όλους τους συναδελφούς από τις πέντε επιτροπές που αντιπροσωπεύτηκαν εδώ και για κάθε επιτροπή έχουμε και πάλι ε, νέα στις 2.30 την κυρία Μπράτουσεκ, την Δευτέρα στις 2.30 και φυσικά θα γίνει η συνεδρία των συντονιστών σήμερα το απόγευμα. Κυρία όμως, ε, η κυρία Βίκη Βόρτα θα σας πληροφορήσει λεπτομερέστερα για τη δική σας επιτροπή. Σε ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή ακόμη. Ε, Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω την κυρία Μπινκόφσκα. Επιζήσατε μέχρι στιγμής, αλλά δεν τέλειωσε. Όχι, καθίστε, δεν χρειάζεται να σηκωθείτε ακόμα. Πρέπει να, να περάσετε και από τη διαδικασία της αξιολόγησης με επιτυχία. Εμείς είμαστε πολιτικοί, δεν ε, συμφωνούμε σε όλα μεταξύ μας. Αν συμφωνούσαμε θα ήταν αλλιώς η ζωή, αλλά τώρα πρέπει να συνεδριάσουμε για να αποφασίσουμε κατά πόσον ε, υπάρχει πλειοψηφία ε, που θα σας ε, κρίνει κατάλληλη για το αξίωμα της Επιτρόπου. Να υπενθυμίσω στις πολιτικές ομάδες ότι αν δεν στείλουν εκπρόσωπο της ομάδας τους ως συντονιστής στις επόμενες ε, συνεδριάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη οι ψήφοι τους, δεν θα καταμετρηθούν στην αξιολόγηση. Είναι σημαντικό λοιπόν για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Λοιπόν, οι συντονιστές της εσωτερικής αγοράς συνεδριάζουν τώρα και κλεισμένων των θυρών η ΙΤΡΕ 6 και 7,5 6 έως 7,5 στο 5G3 και στις 7 η ΙΤΡΕ και η ΙΜΚΟ, συντονιστές πάντα, στην αίθουσα 5G3. Και βέβαια οι εκπρόσωποι και των συνδεδεμένων επιτροπών μπορούν να έρθουν στην τελευταία αυτή συνεδρίαση. Τώρα λοιπόν αυτό που θα γίνει θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ των δημοκρατικά εκλεγμένων συναδέλφων. Ευχαριστώ.